Ε, να συμπεριληφθούν σε επιτροπές ε, και αντιπροσωπείες, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Περιπολισμού κ. Άβελ, ε, στη θέση του κ. Κοζανίνο. Στην Επιτροπή Αναφορών η κυρία Τέιλορ δεν είναι τακτικό μέλος πια. Στην αντιπροσωπεία της συνεργασίας με το Καζακστάν, Κυργιστάν, Ουσμπεκιστάν, σχέσεις Τουρκμενιστάν, Ταζικιστάν, Μογγολία, ο Μισελ Νταντά αντικαθιστά τον κύριο Τσάμπα έρι σχέσεις ε, με την Ουτεαντολική Ασία. Ο κύριος Έρη αντικαθιστά τον κύριο Νταντά, αντιπροσωπεία της Μικτής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας με τη Χιλή. Η κυρία Ιργκοέν Πέρες αντικαθιστά την κυρία Ντεουρκίθα. Η κυρία Νικόλ Σενκλέρ τον Σόσα Βάγνερ στις ε, σχέσεις με την κοινότητα των Άνδεων. Η κυρία Ορκίθα αντικαθιστά την κυρία Ιργόεν Πέρε, την αντιπροσωπεία τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωση για τη Μεσόγειο, ο κύριο Όμπερ Μάγερ στι σχέσει με την Ινδία, κυρία Κριστίνα Μορβάη, την αντιπροσωπεία για τη σχέση με τη ΣΥΠΑ, ο κύριο Τρέβορ Κόλμα, αντικαθιστά την κυρία Κριστίν Μορβάη, για τι σχέσει με την Νότια Αφρική, ο κύριο Βαντερστούμπ, για την ε, Eurolat, Νικόλη Σενκλέρα, αντικαθιστά τον Φρανσίσκο Σόσα Βάγνερ για τις σχέσεις με την Ελβετία και την Νορβηγία και την Ισλανδία και για τον ΕΟΧ, κυρία Σιλβάνα Κοχμερίν. Για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, κυρία Μαρία Λένα Κοπάντη, καθώς τον κύριο Δανέλη. Με το Μεξικό, ο κύριος Φρανσίσκο Σόσα Βάγνερ και για τις σχέσεις με την Ιαπωνία, κύριος Μαγνάντρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, αμέριστη προσοχή σας και ζητώ να μου πείτε αν υπάρχουν ενστάσεις. Ο κύριος Γέμεκ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Στο 323 έδρανο, κύριε Γκέμεκ, δεν θέλετε το λόγο τελικά. Ωραία. Άρα, αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνονται οι ορισμοί αυτοί και περνάμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Θα είμαι πάρα πολύ αυστήρη με το χρόνο αγόρευσης. Μιράντα, για ένα λεπτό, για την έκθεση δεν παρευρίσκεται. Περνάμε στην κυρία Σουίνμπερν. Ένα λεπτό.